Buenas tardes. σας απόγευμα. Να ξεκινήσουμε τώρα την τρίτη στρογγυλή τράπεζα. Θα αλλάξουμε τώρα βέβαια κάπως το πεδίο, διότι εμείς θα συζητήσουμε το θέμα της ενίσχυσης της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, ε, θα ξεκινήσω εγώ δίνοντας το καλό παράδειγμα και θα είμαι πολύ σύντομος στην εισαγωγή μου. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους όσους βρίσκονται εδώ και ιδιαίτερα τον Επίτροπο Κίντ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνο για το θέμα που θα εξεταστεί σήμερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας καλωσορίζω σε αυτή, το, σε αυτή τη συζήτηση. Αυτή η διάσκεψη αναμεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο και οι ε, παρεμβάσεις των ομιλητών ε, θα καταγραφούν. Να σας πω επίσης ότι σήμερα το απόγευμα υπάρχει διερμηνία σε μια σειρά από γλώσσες μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά. Μπορείτε και να μιλήσετε και να ακούσετε ελληνικά. Ο πρόεδρος απαριθμεί τις υπόλοιπες γλώσσες. Σήμερα λοιπόν ε, θα συλλέξουμε μια σειρά από μαρτυρίες. Ο χρόνος για τις παρεμβάσεις δυστυχώς ε, θα είναι 1,5 λεπτό και για τους ε, εμπειρογνώμονες 5 λεπτά θα δώσουμε στον Επίτροπο και 2 λεπτά στους υπεύθυνους, στους εκπροσώπους των διαφορών υπηρεσιών. οι ευρωβουλευτές και τα κράτη-μέλη θα έχουν ένα χρόνο ε, παρέμβασης 1,5 ε, λεπτά. Λοιπόν, η εισαγωγή μου πρώτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Ταγιάννη για την πολύ καλή αυτή ιδέα να οργανωθεί αυτή η διάσκεψη ψηλού επίπεδου και αυτά τα τρία ενημερωτικά πάνελ θα μπω άμεσα στην ουσία του συστήματος. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι σε κάποιο βαθμό έχει μειωθεί η ασφάλεια των συμπολιτών μας. Έχουμε άμεσες ε, αποδείξεις 11 τρομοκρατικές επιθέσεις τις 11 τελευταίες εβδομάδες. Τελευταία χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε και βεβαίως εδώ αναφέρομαι στα κράτη-μέλη εκείνα, στα ε, θεσμικά όργανα, ε, στις υπηρεσίες που ασχολούνται με την ασφάλεια, στις περιφέρειες και στους δήμους. Το δικαίωμα ε, ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η θεμέλια λίθος, ε, θεμέλιος λίθος ε, της ευρωπαϊκής ηθαγένειας και δεν μπορούμε ε, να το εγκαταλείψουμε αυτό. Το 1992 στο Μάστριχτ καταργήσαμε τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Εναρμονίσαμε τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Ε, η ευρωπαϊκή πολιτική θεωρήσεων, η κοινή, ε, ξεκίνησε. Σπουδαία πρόταση. Αστυνομική και δικαστική συνεργασία θέσπιση και ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφοριών Σέγγεν. Αυτή όμως η επιτυχία αυτή τη στιγμή απειλείται, διότι είναι δύσκολο να εντοπιστεί η είσοδος, οι μετακινήσεις ε, και οι πράξεις των τρομοκρατών στο έδαφος της Σέγγεν. Βεβαίως αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να περιορίσουμε τις ελευθερίες που έχουμε κατακτήσει. Βεβαίως πρέπει όλοι μαζί να βελτιώσουμε το σύστημα, να ενισχύσουμε την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης. Και αυτό ακριβώς ε, είναι ο, ρόλος που έχει να λάβει ο Επίτροπος με αφοσίωση και επιτυχία. Πρώτα απ' όλα βέβαια θα πρέπει να εντοπίσουμε τον έστραυστο, τα, τα ευάλωτα σημεία μάλλον. Η πρόσφατη ανακοίνωση της Κομισιόν για την πρόοδο προς μια Ένωση ασφάλεια και αποτελεσματικότητα είναι ένα πρώτο βήμα. Έχουμε εντοπίσει μια σειρά από διαθρωτικέ αδυναμίε που έχουν κάνει μέρο των πληροφορία. Αναφερθώ σε κάποιε από αυτέ. Κενά ενημέρωση ε, και πληροφόρηση ό,τι αφορά τη διαχείριση δεδομένων. Ένα περίπλοκο τοπίο συστημάτων πληροφοριών που λειτουργούν ξεχωριστά. Κατακαιρματισμένη διαχείριση δεδομένων για τα σύνορα και την ασφάλεια όπου αποθηκεύονται ξεχωριστά τα στοιχεία σε συστήματα τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και αυτό μας οδηγεί σε αδιέξοδα. Για να, να αντιμετωπίσουμε αυτές ε, τις ανεπάρκειες, η Κομισιόν προτείνει παρεμβάσεις σε τρεις τομείς. Πρώτον, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα πλεονέκτημα των συστημάτων πληροφοριών που έχουμε ήδη. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε το ΣΥΣ, αλλά και την βάση δεδομένων για το άσυλο ε, και τη Eurodac και το σύστημα πληροφοριών για τα ποινικά μητρώα, το ECRIS. Θα πρέπει επίση να ανοιχτήσουμε την EU Θα πρέπει να δώσουμε νέε αρμοδιότητε στην EU Θα πρέπει να τη δώσουμε και μεγαλύτερο προπολογισμό. Οι εναλλακτικέ για νέε συμπληρωματικέ δράσει για να αντιμετωπίσουμε τα κενά στη δομή τη Ένωση ό,τι αφορά τη διαχείριση δεδομένων τώρα. Ε, έχουμε εντοπίσει σημαντικά κενά σε ό,τι αφορά του υπηκόου τρίτων χωρών που επισκέπτονται τον χώρο Σέγγεν. Εγώ είμαι εισηγητή στην έκθεση για την είσοδο και την έξοδο. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια διαθεσμική συμφωνία πριν το τέλος του μήνα. Εργαζόμαστε σκληρά στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ε, προγράμματος καταγραφής ταξιδιωτικών μετακινήσεων, το αιτία. Επίση υπάρχει το θέμα τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφορία. Δεν πρόκειται τώρα να το αναπτύξω περαιτέρω αυτό, διότι σίγουρα θα το κάνει ο Επίτροπο. Θα πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν τη διαλειτουργικότητα. Και τέλο, και με αυτό κλείνω, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν ε, οι απειλέ του οργανωμένου εγκλήματο που έχει εντοπίσει η Europol στα πλαίσια του ΣΟΚΤΑ. Κυβερνοέγκλημα παραγωγή και εμπόριο ναρκωτικών, διακίνηση προσώπων, οργανωμένο έγκλημα κατά της διοκτησίας, διακίνηση, ε, ε, ε, μάλλον δουλεία, εξέπλημα χρήματος, ε, παραχάραξη και επιγραμμικό εμπόριο παράνομων προϊόντων και υπηρεσιών. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο. Παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που απευθύνατε για τη σημερινή συνεδρίαση. Θα αναφερθώ στα, θέματα, που μου ζητήσατε να θίξω, όμως κάποια πράγματα πρώτα. Όπως είπατε, υπήρξε μια σειρά επιθέσεων, πέντε τον αριθμό του τελευταίο μήνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι σίγουρα θέλουμε να συλληπιθούμε τα θύματα και τις οικογένειές τους. Δεύτερον, χαιρετίζω τη σημερινή σε διάταξη και αυτό το πρόγραμμα, όμως όλοι συμφωνούμε ότι η μετανάστευση και η ασφάλεια έχουν ξεχωριστές προκλήσεις και δεν θα πρέπει να συγχέονται ως ένα και το αυτό ζήτημα. Είναι ένα προπέτασμα που συχνά αξιοποιούν λαϊκιστές και εξτρεμιστές. Τρίτον, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ 100% με τους προηγούμενους ομιλητές της προηγούμενης συνεδρίασης που είπαν ότι η αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική ε, που θεμελιώνεται στο σεβασμό προς τις ε, θεμελιώδεις αξίες μας και αρχές μας είναι βασικό ε, κλειδί στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και του ακραίου εξτρεμισμού και έτσι διασφαλίζουν και την ασφάλεια σε όλα τα κράτη-μέλη. Όμως ένα βασικό σημείο είναι και η ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά μας σύνορα αλλά και η ενίσχυση της ε, ασφάλειας και της συνεργασίας εντός των σύνορων. Στα εξωτερικά μας σύνορα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της προστασίας, συλλογικής προστασίας, από κοινού δηλαδή των κοινών μας σύνορων και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα στηρίξουμε. Τον περασμένο Οκτώβριο δημιουργήθηκε η συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή. Ακούσαμε ήδη από τον κύριο Λετζέρη για τη δουλειά ε, που επιτελεί και τους τελευταίους μήνες έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και πλέον ε, έχει σημαντικό αριθμό συνοριοφυλάκων σε διάφορα σημεία, σε, όλα, ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα εξωτερικά της σύνορα δηλαδή, συμπληρώνοντας τις υφιστάμενες δομές σε ό,τι αφορά τη συνοριοφυλακή. Για την ασφάλεια, πέραν τη στήριξη ε, προ ε, τα κράτη-μέλη και την επιστροφή των παράνομων μεταναστών, ο οργανισμός ε, παρέχει αρρωγή στα κράτη-μέλη στον τομέα τη πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματο. Και έχουμε δει όλοι τι συμβαίνει με του αλλοδαπού μαχητέ που προσπαθούν να επισέλθουν στι στις μεταναστών. Έχουμε ενισχύσει τους ελέγχους στα hot spots στην Ελλάδα και στην Ιταλία Έχουμε προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, αλλά και από την Europol, για να στηρίξουμε τις εθνικές αρχές. Γενικώ, όπω ε, ανέφερε και ο Πρόεδρο, έχουμε ενισχύσει ε, τα όσα γνωρίζουμε για αυτού που εισέρχονται και εξέρχονται των συνόρων μα, των εξωτερικών συνόρων, με την αναθεώρηση του κώδικα Σέγγεν. Όλοι όσοι εισέρχονται και εξέρχονται τη Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά ελέγχονται στο σύστημα SIS, που είναι η πιο σημαντική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς επιβολής του νόμου. Όπως ανέφερε και πάλι ο Πρόεδρος, η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου μεταναστών ε, απαιτεί διασυνορική συνεργασία μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών με τη στήριξη και του αρμοδίου κέντρου στη Europol και είναι εδώ και ο διευθυντής Μαρτίνο προσωπώντα τη Europol και θα σα τα πει στη συνέχεια. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μα με τρίτες χώρε. Τον Ιανουάριο η Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση για την οδό τη Κεντρική Μεσογείου που αναφέρει μια σειρά ε, μεθόδων συνεργασία ε, με τρίτε χώρε που θα μα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση ε, τη διακίνηση και η επιχείρηση Σοφία έχει ήδη αναφερθεί σήμερα το απόγευμα ε, με μια ανεπιτυχή αντιμετώπιση των διακινητών και χαίρομαι που ε, είναι εδώ και ο ε, συνάδελφος που μας θα πει στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές, μια σειρά των μελών επανεσύγαγαν προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους. Στις αρχές της χρονιάς η Επιτροπή συνέστησε αυτή η έλεγχη να αρθούν προκειμένου να βοηθήσουμε τα κρατημέλη στη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων, παρουσιάσαμε ε, μέτρα για να ενισχύσουμε τους αστυνομικούς ελέγχους και την αστυνομική συνεργασία όπου δει ε, σε όλο το χώρο Σέγγεν έως και τις ε, συνοριακές περιοχές. Ενθαρρύνουμε επίσης τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία μέσω κοινών περιπολιών της αστυνομίας, διασυνοριακούς ελέγχους, κοινή ανάλυση κινδύνου και απειλών ε, και ενισχυμένη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών. Και μάλιστα η ανταλλαγή πληροφοριών αυτή, αν ενισχύσουμε δηλαδή τη συνεργασία μας μεταξύ των κρατών μελών, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για να αυξήσουμε και τα επίπεδα ασφάλειας. Απαιτούνται λοιπόν ανταλλαγές πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ κρατών μελών, ενωσιακών οργανισμών, επιβολή του νόμου και ε, δικαστικές αρχές, αλλά και μυστικές υπηρεσίες. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα νομοθετικών μέσων και συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών για να διευκολύνουμε ακριβώς ε, αυτή τη συνεργασία μεταξύ των ε, αρχών. Έχουμε το SIS, το VIS, το δίκτυο Broom, το Σύντομα θα έχουμε και την οδηγία ε, για τα στοιχεία των ταξιδιωτών, το NPR, και η πρόσφατη οδηγία καταπολέμησης θερμοκρατία που ενισχύει το νομοθετικό πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών για, τις, για σκοπούς ε, καταπολέμησης θερμοκρατίας. Οι ευρωπαϊκοί μας οργανισμοί, πιο συγκεκριμένα η Europol, διαδραματίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην διευκόλυνση της ε, ανταλλαγής πληροφοριών. Του των αναπόφευκτα και αναμφίβολα υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Έχουμε κάνει μια σειρά προτάσεων, είτε για να ε, ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε την ε, λειτουργία εφιστάμενων δομών, είτε για να καλύψουμε τυχόν κενά προτείναμε την ενίσχυση του ε, συστήματο ανταλλαγή προφοριών Schengen ε, βάσει τη υφιστάμενη εμπειρία. Οι προτάσει που κάναμε έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν την ανταλλαγή προφοριών σε όλη την Ευρώπη σε σχέση με την τρομοκρατία ε, και να αυξήσουμε την χρήση ε, των βιομετρικών στοιχείων. Θεωρούμε ότι έτσι θα βοηθήσουμε τους αξιωματούχους που ενεργούν στα εξωτερικά σύνορα και χαίρομαι ιδιαίτερω που ο εισηγητή ε, σε αυτόν τον σημαντικό φάκελο Κοινοβουλίου θα συμμετάσχει σήμερα στη συζήτηση. Η υιοθέτηση και υλοποίηση του συστήματος εισόδου-εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΕΤΙΑΣ, το αντίστοιχο ανάλογο σύστημα ΕΣΤΕΡ ε, των ΗΠΑ, θα μας βοηθήσει να ξέρουμε καλύτερα ποιος μπαίνει και βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, που βαίνουν καλώ ε, οι διαπραγματεύσει και ευχαριστώ τον Πρόεδρο για όλε τι προσπαθίε του σε αυτό το σημαντικό φάκελο και ελπίζω όντω να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, όπω είπε και ο ίδιο. Θα εξετάσω το αίτια μαζί με κάποιου από εσά και γιατί είναι σημαντικό για την εσωτερική μα ασφάλεια και για το μέλλον τη ε, πολιτική θεωρήσεών μα. Και επί τη ευκαιρία και πάλι να σα παροτρύνω όλου ε, να μα βοηθήσετε να καταστήσουμε επιχειρησιακό το αίτημα αίτιας το στομότερο δυνατόν. Δύο λόγια τώρα για αυτό το ζήτημα της ε, Έχουμε συστήσει μία ομάδα προγνωμόνων για τα πληροφοριακά συστήματα και την ε, διαλειτουργικότητα, ακριβώς για να εξετάσουμε τις επιμέρους επιλογές που υπάρχουν, ε, ούτω ώστε τα πληροφοριακά μα συστήματα να συντονίζονται με καλύτερο τρόπο και έτσι ε, να καλύψουμε ορισμένα κενά που υπάρχουν. Η ομάδα ε, κατέληξε σε κάποιες συστάσεις στις αρχές χρονιάς και πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι προτάσεις για μια ευρωπαϊκή κοινή διαπαφή, ένας ε, κοινός χάρτης ε, βιομετρικών στοιχείων και ένα αποθετήριο ε, ήταν ε, εφικτές λύσεις που θα μπορούσαν να μας δώσουν ε, απτά αποτελέσματα σε πλήρη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις και τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει αυτά τα ευρήματα και πρότεινε ε, και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Πρέπει αρχικά να συνεργαστούμε, να από κοινού για να κλείσουμε όλους τους εκκρεμείς φακέλους που αφορούν ακριβώς ε, τα συστήματα ανταλλαγή προφοριών. Την επόμενη εβδομάδα θα υποβάλουμε μέτρα για την ενίσχυση του EU Lisa και βλέπω ότι ο διευθυντή είναι εδώ μαζί μας και θέλουμε και να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό ε, Σύστημα Ποινικού Μητρώου που αναφέρατε και στις Πρόεδρε. Ταυτόχρονα θέλουμε μαζί με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουμε σε μια κοινή θεώρηση των απαραίτητων βημάτων για να επιτύχουμε την διαλειτουργικότητα αυτή. Να κλείσουμε λοιπόν τα εκκρεμή ζητήματα και μαζί με αυτό που προανέφερα θα μας φέρει ε, σε ένα στάδιο όπου θα μπορέσουμε να υποβάλουμε προτάσεις, νομοθετικές προτάσεις στις αρχές του 2018 για αυτό το ζήτημα. Κυρίες και κύριοι, για να διασφαλίσουμε αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ε, την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας κοινό μας στόχος και πρέπει να συνεχίσουμε την κοινή αυτή προσπάθεια. Προσβλέπω στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας και σήμερα και στις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ευχαριστώ. Σα σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε, για τα λόγια σας, που είναι πάντα έξυπνα και πάντα αποφασιστικά ο μεγάλος ειδικό ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα του Σέγγεν, ο κύριος Κάρλος Κοέγιο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Η πολιτική ασύλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα τεράστιο θέμα. Χρειαζόμαστε συντονισμένες δράσεις για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις της ασφάλειας και της μετανάστευσης. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό χρόνο ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ορισμένοι λένε ότι έχει καταρρεύσει το Σέγγεν. Το Σέγγεν θα πρέπει να είναι η λύση και για την τρομοκρατία και για την ασφάλεια. Θα πρέπει να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα, να προωθήσουμε την νομοθεσία, να συντονίσουμε τη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σύστημα ε, ε, πληροφόρησης του Σέγγεν, το ΣΥΣ, είναι το μεγαλύτερο σύστημα πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρησιμοποιείται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Συνεισφέρει στην ασφάλειά μας. Με το ΣΥΣ πρέπει να έχουμε καλύτερη συνεργασία και καλύτερη ενημέρωση μέσω των νέων συστημάτων καταχώρησης. Το ΣΥΣ μα δίνει και νέα εργαλεία για την καταπολέμηση τη δημοκρατία και τη σοβαρή εγκληματικότητα με περισσότερε βιομετρικέ πληροφορίε και την υποχρέωση επιμερισμού των πληροφοριών για την τρομοκρατία και του ξένου μαχητέ. Το ΣΥΣ θα έχει και νέα εργαλεία για να δώσει απαντήσει στην κρίση τη μετανάστευση, εξασφαλίζοντα την πρόσβαση στα hot spot. Το ΣΥΣ θα προστατεύσει κυρίως τα παιδιά, δημιουργώντας συστήματα ενημέρωσης και έγκαιρης προειδοποίησης. Το ΣΥΣ επιτρέπει τον επιμερισμό των πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και τη βοήθεια για μια αυξημένη ε, συνεργασία. Η αποτελεσματικότητά μας εξαρτάται από το ΣΥΣ για να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, για να διασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια των πολιτών, δεν πρέπει να επανεφεύρουμε τον τροχό πρόεδρε. Θα πρέπει να χτίσουμε πάνω στις βάσεις που διαθέτουμε ήδη, με συστηματικό και προγραμματισμένο τρόπο. Ελπίζω ότι οι μελλοντικέ εργασίες μας, ειδικά σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφορικής και ενημέρωσης, να ακολουθήσει αυτό το μοντέλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κάρλος που είπες τόσα σημαντικά πράγματα σε τόσο λίγο χρόνο. Και τώρα, το λόγο έχει μία ε, δήμαρχος από την Ουγγαρία, η Άννα Μαχιάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δώσατε το λόγο. Εκπροσωπώ μία περιοχή κοντά στα σερβικά σύνορα, στα σύνορα Σέγγεν. Ξέρουμε ότι οι ανθρωπιστικές πτυχές ε, του θέματος αυτού θα πρέπει να ειδωθούν σε συνδυασμό με τα δικαιώματα και την κατάσταση την οποία βιώνουν οι ίδιοι μας οι πολίτες. Είδαμε ότι μόνο λίγοι από αυτούς που περνάνε παράνομα τα σύνορα το κάνουν γιατί πραγματικά χρειάζονται βοήθεια. Πολλοί έρχονται χωρίς έγγραφα. Και είχαν και iPhone. Λίγο περίεργο, έτσι και έρχονται από παραπάνω από 100 χώρες. Δεν υπάρχουν πόλεμοι σε 100 χώρες παρόλα αυτά. Οι περισσότεροι έρχονται από το Πακιστάν και τον Μπαγκλαντές. Ο κόσμος στην περιοχή μου θέλει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των πραγματικών προσφύγων και όχι των, των οικονομικών μεταναστών. Είναι μια κυρίαρχη απόφαση της χώρας μου να αποφασίσει ποιος γίνεται δεκτός και ποιος όχι. Είναι υποχρέωση της Ουγγαρίας να υπερασπιστεί τα σύνορα Σέγγεν, τα σύνορά της με τη Σερβία δηλαδή. Πρέπει να παρεμποδίσουμε την παράνομη διέλευση των σύνορων αυτών. Και με αυτόν τον τρόπο αν το κάνουμε αυτό, θα προστατεύσουμε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο η Ουγγαρία βοηθάει για να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση. Θα θέλαμε αυτό να αναγνωριστεί. Γιατί είναι σημαντικό. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να μας ε, δώσει ένα μήνυμα αλληλεγγύης η πόλη των Βρυξελών. σα ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Και τώρα το λόγο έχει ο υποδιευθυντής της Europol, ο κ. Μαρτίν. Thank Πρόεδρε, ευχαριστώ και καλησπέρα. Θα ήθελα, εν συντομία, να συμπληρώσω και να υποστηρίξω κάποιες από τις παρατηρήσεις του Επιτρόπου κυρίου Κίνγκ. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια δεδομένη δραστηριότητα οργανωμένου εγκλήματος που ωστόσο δείχνει ότι υπάρχει μια οργανωμένη αγορά με κέρδη έως και 3 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση τις εκτιμήσεις μας και δραστηριότητες και σε άλλους τομείς εγκληματικής δραστηριότητες με χαμηλό κίνδυνο. Ενώ για τους ίδιους, για τα θύματα αυτών των δικτύων ε, μετανάστες και παιδιά. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος και με πολύ αριθμούς θανάτους, Γι' αυτούς ο κίνδυνος είναι μηδενικός. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ε, προηγμένη και θα ήθελα εγώ να σας εκθέσω εδώ ποιος είναι ο ρόλος της όλο, όταν εξετάζουμε τις δραστηριότητε που μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο για τον ε, λάθρο διακινητή και να περιορίσουν και τα το κέρδος από τη δραστηριότητά του αυτή. Έτσι λοιπόν έχουμε θεσπίσει ένα κέντρο εδώ και ένα χρόνο, κέντρο διακίνησης ε, μεταναστών. Έχουμε συνεργασία με τη Frontex, την EASO, την ε, UNAF, την Interpol και άλλους κύριους παράγοντες και φορείς. Έχουμε ε, διάφορες επαφές σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία και δευτερογενείς ελέγχους για την διάγνωση πιθανού κινδύνου για ε, τρομοκρατική δράση. Ενισχύουμε τη διασυνοριακή συνεργασία. Περί τις 50.000 είναι οι διακινητές που έχουμε καταγράψει στη βάση δεδομένων μας και έχουμε υποστήριξη διαγραμμική 60 διαφορετικών επιχειρήσεων. Έχουμε προχωρήσει διάγνωση 2.000 διαφορετικών υποθέσεων στο κέντρο για τους μετανάστες έχουμε 46, κυρίως σε πρωτεύουσε αυτή τη στιγμή. Για το μέλλον τώρα, θέλω να τονίσω ιδιαίτερα την διαλειτουργικότητα και την επανεξέταση του τρόπου ε, συνεργασίας, ανάπτυξης της βάσης δεδομένων και τη δίωξη των διακινητών. Ως παράδειγμα, θέλω ιδιαίτερως να τονίσω τη πρόσφατη εξέλιξη στο Eurodac με την ανάπτυξη μιας μονάδας για τους ανήλικους, υπάρχουν θύματα της διακίνησης, και επίσης ως ε, εκδήλωση στήριξη στη διακήρυξη της Μάλτας έχουμε αναλάβει νέα καθήκοντα κυρίως ανταλλαγή δεδομένων με διάφορους παράγοντες, τρίτους ε, με στρατιωτική αλλά και αστυνομική, με αστυνομικές αλλά και στρατιωτικές δομές και ενισχυμένη εστίαση στις συνεργατικές δράσεις με τις αποστολές της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας που μπορούν να φέρουν σημαντικά επιχειρησιακά ωφέλη. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αυτά τα νέα καθήκοντα. Χρειάζονται όμως επιπλέον πόροι οι τρέχουσες προβλέψεις, οι δημοσιονομικές, δεν μας εξασφαλίζουν τους απαραίτητους πόρους. Θέλω ωστόσο να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και τους λοιπούς θεσμούς και φορείς που μας έχουν υποστηρίξει. Σας ευχαριστώ και εγώ. Διαβιβάστε τις, τους χαιρετισμούς μου στον διευθυντή σας, τον κύριο Ρόμπα. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Φαμπρίς Λεζερή, που είναι ο πρόεδρος της Frontex. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, ε, υποδοχή σας και θα ήθελα να πω, όπως ακούστηκε και νωρίτερα, ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην ασφάλεια των εξωτερικών μας συνόρων με τη συνεργασία αυτή και θέλω ιδιαίτερα δύο μηνύματα να διατυπώσω ότι με τη νέα εντολή έχουμε καταστεί παραγόντες διαμόρφωσης της πολιτικής ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να συνεργαζόμαστε και με τις δυνάμεις του νόμου, την αστυνομική την δυνάμεις αλλά και την Europol με νέες δυνατότητες για συλλογή προσωπικών δεδομένων στη διάρκεια των κοινών μας επιχειρήσεων, ε, της ε, ανάπτυξης των δυνάμεών μας, τα εξωτερικά σύνορα μπορούμε να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, τα οποία μπορούν να διατεθούν και διατίθενται στη Europol, τις τοπικές αστυνομικές αρχές και που συμβάλλουν ε, στις αστυνομικές έρευνες και στη δίωξη του εγκλήματος ιδιαίτερα. Συμβάλλουμε στην τελωνιακή συνεργασία επίσης, και πρέπει να αναπτύξουμε και κάποιες ε, δραστηριότητες ακτοφυλακής. Υπάρχει λοιπόν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπου η Frontex πιστεύω μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα με τους εταίρους και να συμβάλλει περισσότερο στην καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων και την μετατροπή των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα είδος δικού δικτύου ασφαλείας, για τη διαφύλαξη τη εσωτερική ασφάλεια και των συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Για την διαλειτουργικότητα, μια παρατήρηση, τα πράγματα βαίνουν καλώ και θα ήθελα να πω ότι ε, το πόρταλ, ε, η θηρίδα για την ενιαία ε, έρευνα, ε, που ανακοινώθηκε νωρίτερα έχει προχωρήσει. Ήδη έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Ιουλίζα και την Europol αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι η εξασφάλιση πρόσβασης για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες στα προσωπικά δεδομένα είναι μια σωστή επιλογή που μπορεί και να στηρίξει τα κράτη-μέλη στις προσπαθίες τους και να εξασφαλίσει την εσωτερική ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την προσπάθεια λακωνικότητας. Η κυρία Κατερίνα Κινίτσι, που είναι και φίλη μου, έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το θέμα της μετανάστευσης και της ασφάλειας είναι οι πιο σημαντικές και οι πιο δύσκολες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, και με την εξασφάλιση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα. Ε, είδαμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις που ε, διέπραξαν ε, Ευρωπαίοι πολίτες ε, που επέστρεψαν από ζώνες μαχών. Δεν αποκλείεται διάφοροι τέτοιοι ξένοι μαχητές να μεταμφιεστούν ως τούντες άσυλο ή μετανάστες και να μπουν μέσω των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα, σύνορα του Σέγγεν, ώστε να εξασφαλίσουμε την επιβίωση του χώρου Σέγγεν και έλεγχοι που πρέπει να γίνονται πάντα χωρίς προκλήσεις, χωρίς δυσαναλογίες, χωρίς να παρεμποδίσουμε την ελευθερία μετακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών. Χρειάζεται επίσης συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ε, που βοηθιέται και με την ανταλλαγή δεδομένων μέσω των καταλήλων βάσεων δεδομένων. Το σύστημα N36, το σύστημα αιτία, επί των οποίων ε, εργαζόμαστε, είναι πολύ σημαντικά. Τα κράτη-μέλη όμω θα πρέπει να έχουν και νέα συστήματα ανταλλαγή πληροφοριών, το PNR α πούμε, και να χρησιμοποιούν 100% τα ισχύοντα συστήματα μέχρι να εξασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική διαλειτουργικότητα. Τελευταίο, υπάρχει ένα θέμα επί του οποίου πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Είναι το θέμα που αφορά την καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων που διαχειρίζονται τη διακίνηση ανθρώπων, κυρίω στη Μεσόγειο. Δεν είναι αποδεκτό άτομα τα οποία φεύγουν από περιοχές σύγκρουση, από πολέμους, από διώξει, από μια ζωή που δεν έχει καμία αξιοπρέπεια, να πρέπει να πέφτουν στα χέρια των ανθρώπων αυτών που τους εκμεταλλεύονται, που παραβιάζουν τα δικαιώματά τους, κυρίως παραβίαση τα δικαιώματα γυναικών και παιδιών. Πρέπει να παρέμβουμε με πιο αποτελεσματικά εργαλεία. Αυτό σημαίνει επίση καταπολέμηση και τη τρομοκρατίας που χρηματοδοτείται συχνά μέσω αυτή τη διακίνηση ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Ο Ηλίας Στάθης από τον ε, από το γραφείο του ΟΗΕ υπεύθυνο για τα ναρκωτικά και το έγκλημα. Ευχαριστώ, κύριε και κύριοι. Εμείς λέμε ότι χρειαζόμαστε ένα δίκτυο για να καταπολεμήσουμε τις σπήρες των εγκληματιών και πρέπει να βασιστούμε σε μια κοινή κατανόηση για το τι είναι ε, ακριβώς η διακίνηση και πώς επωφελούνται οικονομικά τα δίκτυα αυτές τις σπήρες. Έχουμε προσυπογράψει το πρωτόκολλο της σύμβαση μάλλον ε, και έτσι έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο και έχουμε δώσει τα απαραίτητα εφόδια στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Όμως, ε, οι ε, δίωδοι διακίνηση ε, δεν αφορούν μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι πρέπει να διευρύνουμε τις προσπάθειές μας για να εντοπίσουμε ακριβώς αυτέ τι πύρε όπου συλλέγονται τα χρήματα τα μέσα ε, συνεργασία αυτών των κοινών διόδων, ακόμα και χωρίς διμερεί συμφωνίες υπάρχουν και η Σύμβαση του Παλέρμου αυτό μα ε, επιτρέπει. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ε, το φαινόμενο αυτό από τις οργανωμένε εγκληματικέ πύρες. Ε, το κέρδο είναι κεντρικό χαρακτηριστικό του αδικήματος αυτού και αυτό καλούμε όλους του ενδιαφερόμενους φορεί να ακολουθήσουν και να εκμεταλλευτούν τα χρήματα να δεσμεύσουν ε, πόρους που συνδέονται με αυτή την παράνομη δραστηριότητα. Πρέπει περισσότερες προσπάθειες να καταβληθούν και στην Ευρώπη και ευρύτερα ε, για την αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων μέσω συγκέντρωσης ε, πληροφοριών και ανταλλαγής πληροφοριών. Να ακολουθήσουμε λοιπόν τα χρήματα μαζί με μέτρα κατά τη διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Εγώ σα ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Η ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης είναι, πιστεύω, ένα σημείο που συμφωνούμε όλοι. Όσο αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση, αυξάνονται και τα επίπεδα των απειλών που αντιμετωπίζουμε, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την τρομοκρατία. Αυτό κατέδειξαν άλλωστε τα τελευταία γεγονότα. Ω εκ τούτου, είναι πολύ σημαντική η αποτελεσματική και ουσιαστική χρήση ποιοτικών πληροφοριών. Οι υπηρεσίε ασφαλείας και οι συνοριοφύλακε είναι κρίσιμη κρίκη στην αλυσίδα του έγκαιρου εντοπισμού πιθανών πηγών κινδύνου και αποτελεσματική αντιμετώπιση. Η χρήση τη τεχνολογία, η ενοποίηση των συστημάτων, τα κράτη-μέλη να επικοινωνούν μεταξύ του με ένα σύστημα είναι πολύ σημαντικό στην καταπολέμηση αυτού του κινδύνου. Χρειάζεται επίση να βρούμε του τρόπου για να συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια και οι εταιρείε τεχνολογία. Ακούσαμε πριν για την χρήση των μέσων κοινωνική δικτύωση, οι κολοσσοί των οποίων συντονίζονται οι τρομοκράτε. Χρειάζεται όμω να βρούμε και την ισορροπία. Οι βασικέ αρχέ λειτουργία τη Ένωση είναι ακρογωνιαίο λήθο. Η ελευθερία διακίνηση δεν πρέπει να καταπατηθεί στην προσπάθεια ενίσχυση των ελέγχων στον χώρο Σέγγεν. Σε αυτό το πλαίσιο στηρίζουμε ως Κύπρος τις πρωτοβουλίες που γίνονται σε νομοθετικό και επιχειρησιακό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το πακέτο των έξυπνων συνόρων, την δημιουργία της ακτοφυλακής και την πρόταση για την παραχώρηση προέγκρισης εισόδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ε, για την αντιμετώπιση της ε, σωματεμπορία. Στην κυρία Μύρια Βασιλιάδου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Ήθελα μόνο να σταθώ πιο συγκεκριμένα στην διακίνηση ανθρώπων στην εμπορία ανθρώπων είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο, αλλά όταν ε, μιλούμε για το οργανωμένο έγκλημα, είναι η μοναδική μορφή οργανωμένου εγκλήματο η οποία εγγράφεται στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ω ένα πολύ σοβαρό ε, αδίκημα, ως πολύ σοβαρή παράβαση. Είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε. Έχουμε ένα ε, ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξωτερική διάσταση είναι στο τμήμα τη πολιτική πολύ πριν ξεκινήσει η μεταναστευτική κρίση. Και έτσι παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις προ... προπαρασκευαστικές εργασίες ε, ε, για τον παγκόσμιο αντίκτυπο της μετανάστευση μέσω ε, με συγκεκριμένη συζήτηση για την εμπορία ανθρώπων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προκλήσεις και αυξημένες απειλές κατά της ασφάλειας που έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε αυτό το φαινόμενο. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Οι τάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι αρκετά σταθερέ τα τελευταία 6-7 χρόνια και η Europol είναι η πιο σημαντική πηγή πληροφόρηση. Τα δύο τρίτα των ε, ε, θυμάτων της διακίνηση ανθρώπων είναι η τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα δύο τρίτα των διακινητών. Και αυτό είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε. Να πω μόνο ότι σε ό,τι φορά την μεταρρυθμιστική κρίση, οι διακινητές αξιοποιούν όλο και περισσότερο την κρίση ε, για να πλήξουν ε, του πλέον ευάλωτους, τις γυναίκε και τα παιδιά. Και να δώσω ένα παράδειγμα εδώ. Ε, ο IOM και η UNICEF λένε ότι αυξανόμενο αριθμό νιγηριανών επικών, γυναικών και παιδιών φτάνουν μέσω Λιβύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 11.000 γυναίκε και παιδιά το 2016, διπλάσιος αριθμό το του 2015. 25 φορές περισσότερο από ότι το 2013. 80% ε, εκτιμάται ότι είναι θύματα διακίνησης ε, ε, ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς κακοποίησης και υπάρχουν σημαντικές παραβάσεις στο το σύστημα ασύλου και ακούμε από ότι αγνοούνται θύματα σεξουαλικής κακοποίησης μετά την αφήξή τους Κάποιοι ενήλικες εμφανίζονται και ζητούν να τους δώσουν ένα ε, παιδί, υποθέτω ότι είναι συγγενείς. Διακόπτε ο Πρόεδρο. Θέλουμε τώρα να τα συνδέσουμε όλα αυτά και με άλλε μορφέ εγκληματικότητα και έχουμε και το ψήφισμα του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ε, που συνδέει ακριβώ τη διακίνηση ανθρώπων με άλλε εγκληματικέ ενέργειε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ ξεκάθαροι γιατί δεν είναι το ίδιο και το αυτό. Και ο Πρόεδρος και η Europol μας είπαν ότι η διακίνηση ανθρώπων είναι προτεραιότητα να καταπολεμηθεί στην ΣΟΚ το 2017. Πρέπει να εξετάσουμε ξεχωριστά την ε, εμπορία ανθρώπων γιατί υπερβαίνει το θέμα ε, της μετανάστευσης. Και κλείνοντας να πω ότι πέραν του μεταναστευτικού φαινομένου πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτό είναι έγκλημα ε, με βάση σημαντικά κέρδη που υπάρχουν και στην νόμιμη και στην ε, μαύρη αγορά. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε τις χρηματικές ροές. 11.000 λοιπόν γυναικόπαιδα από την Ιγυρία, 10.000 ε, κακοποιήσεις κάθε χρόνο, 30 ευρώ ανακακοποίηση, 350 ας πούμε ημέρες τον χρόνο πολλαπλασιάστε το επί 11.000 και έτσι έχετε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Βασιλιάδου, για τη δουλειά σας, πολύ σημαντική δουλειά σας και για τη μαρτυρία σας, πολύ σκληρή. Και τώρα θα δώσω ε, το λόγο στον συνάδελφο από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, στον Gerard Growell. Έχετε το λόγο. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ελληνική και την κάλυψη των προσδοκίων των πολίτων. Θέλω να υπενθυμίσω ότι δεν είναι τρομοκράτης ο κάθε μετανάστης, όπως και ο κάθε μετανάστης δεν είναι ε, μετανάστης. Έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα πολύ συγκεκριμένα στο πρόσφατο παρελθόν. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα για την καταχώρηση των μεταναστών που φτάνουν ε, στις, ε, στα σημεία εισόδου, αλλά δεν μας επιτρέπει κανένα τέτοιο σύστημα να, μας, να, επιλέξουμε ποιον θα, επιτρέψει, θα επιτρέψουμε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επαληθεύοντας δηλαδή ποιο είναι αυτός ο συγκεκριμένο που κάθε ενώπιον του ε, υπαλλήλου που του παίρνει συνέντευξη γιατί ε, έγγραφα ταυτότητα δεν υπάρχουν και φαντάζομαι ότι οι διακινητές τους τα αφαιρούν ή ότι δεν είχαν ούτε καν κατά τη διάρκεια του τέτοια ταξίδια. Φτάνει λοιπόν κάποιο, τον ρωτάνε ποιο το όνομά του, μπορεί να πει όποιο όνομα θέλει, μπορεί να πει όποια χώρα προέλευση θέλει. Άπαξ και μπει μέσα στο σύστημα και καταχωριστεί, τότε είναι ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η ε, ζωή και δραστηριότητά του και αντίστοιχα των αστυνομικών αρχών. Γι' αυτό η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την διακίνηση ανθρώπων. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτό να το εξασφαλίσουμε. Ταυτόχρονα αφήνοντας ε, ένα παράθυρο για την μετανάστευση στην Ευρώπη, χωρίς βέβαια να αρνηθούμε τις ε, πολλές φορές ακραίες ανάγκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών που φτάνουν, που φεύγουν από τον ε, πόλεμο, από σκληρέ συνθήκε και πρέπει να βρουν ένα ασφαλή λιμένα. Ωστόσο υπάρχουν πραγματικά προβλήματα και κάποιο πρέπει επιτέλου να μα δώσει μια απάντηση πώ θα τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Τώρα το λόγο έχει ο Κρούμ Γκάρκοφ, πρόεδρος της EU Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετάσχω στη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική και θέλω να πω στην αρχή ότι σήμερα στην Ευρώπη έχουμε μια διτή πρόκληση να αντιμετωπίσουμε. Από τη μία να παραμείνουμε ανοιχτοί, γιατί όλο και περισσότεροι έρχονται εδώ για να δουλέψουν, να μελε... σπουδάσουν ή να αναζητήσουν προστασία και παράλληλα να παραμείνουμε ασφαλεί, ασφαλείς, να δώσουμε ασφάλεια και προστασία στους Ευρωπαίους πολίτες με σεβασμό παράλληλα των θεμελιακών ε, αξιών και δικαιωμάτων πάνω στα οποία χτίστηκε η Ευρώπη. Η καλύτερη απάντηση λοιπόν γι' αυτό, σε αυτή την πρόκληση, είναι να κρατήσουμε το Σέγγεν, γιατί η ελευθερία μετακίνηση είναι μία από τα μεγαλύτερα, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμή. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε παράλληλα ότι σήμερα η διαχείριση τη μετανάστευση και η εσωτερική ασφάλεια εξαρτώνται απόλυτα από τι πληροφορίε από τη διάθεση και από τη σωστή κυκλοφορία των πληροφοριών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε διάφορα πράγματα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι σημερινέ και αυριανέ προκλήσει. Καταρχά, θα πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλε τι πλευρέ τη, σε όλε τι πτυχέ τη, ούτω ώστε να χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά τα ισχύοντα συστήματα. Και τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό, οι σημαντικέ πρωτοβουλίε όπως το σύστημα εισόδου-εξόδου ή το αιτία θα πρέπει να ενισχυθούν. Θα πρέπει να δουλέψουμε επ' αυτών πολύ πιο σοβαρά, ούτως ώστε να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν και να διευκολύνουν ούτως ώστε να διαχειριστούμε με καλύτερο τρόπο τις ε, μελλοντικέ ε, και σημερινέ ε, μεταναστευτικέ ροές και τις προκλήσεις γενικά. Φυσικά η Ιουλίσα εμπλέκεται σε όλα αυτά. Θα συνεχίσω να εργάζομαι πάνω σε αυτά τα θέματα και με επιπλέον πόρους πιστεύω θα καταφέρουμε να δουλέψουμε επιτυχώς σε όλα τα μέτωπα που θα δώσουν απάντηση στις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο δίνω στο φίλο μου, τον κύριο Μάουρο, Μάουρο, Μάριο Μάουρο. Ε, χαίρομαι που είναι εδώ και που είναι, ε, θα μιλήσει εδώ στο Κοινοβούλιο ο Υπουργό Άμυνα τη ε, Ιταλία. Η Ιταλική Γερουσία δεν έχει πια καμία αμφιβολία μετά από τις έρευνες που έκανε τα τελευταία χρόνια για τους αντικειμενικούς δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των εγκληματικών οργανώσεων, των τρομοκρατικών οργανώσεων και τη διακίνηση των ανθρώπων. Αυτό έχει αποδειχθεί όχι μόνο από τις συλλήψεις που έκανε η αστυνομία της Κατάνια, η εισαγγελία της Κατάνια, το 2013 17 Αιγύπτιοι διακινητές συνελήφθησαν και δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν καθόλου την παρουσία τους. Ε, γιατί κάποια στιγμή βρέθηκαν σε μια περιοχή μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν. Για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Επίσης, στη Λαμπεντούσα το 2011 έφτασε ο, ο δράστης της επίθεσης του Βερολίνου. Πριν από λίγε μήνε, οι Ιταλικές υπηρεσίες ε, συνέλαβαν Κωσοβάρου στη Βενετία, λίγε ώρε πριν από την διάπραξη μια τρομοκρατική επίθεση. Η παρακολούθηση όλου αυτού του περίεργου ε, και περίπλοκου μεταναστευτικού φαινομένου μα λέει, μα αποδεικνύει ότι υπάρχουν δεσμοί, αν ακολουθήσουμε το χρήμα, θα δούμε ότι υπάρχουν δεσμοί όχι μόνο με τι ε, τις εγκληματικές οργανώσεις, αλλά και, με τι τρομοκρατικέ οργανώσει, Δηλαδή διακινητέ, τρομοκρατικέ οργανώσει, εγκληματικέ οργανώσει. Όπως είπε και ο κύριος Κοέλιος στην αρχή της συζήτησής μας, ε, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το αποτελεσματικό κανάλι. Να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι εκ των όνου κάνευ για να καταπολεμήσουμε σοβαρά την τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστώ, Μάριο. Και τώρα το λόγο έχει ένας εκπρόσωπος της επιχείρησης Σοφία, ο Ματέο Σοντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινήσαμε τον Ιούνιο του 2015 στο πλαίσιο τη ευρύτερη ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει μια ολοκληρωμένη απάντηση στη μεταναστευτική κρίση και στο προσφυγικό και να έχουμε μια καλύτερη και πιο ευημερή Λιβύη. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την διακίνηση ανθρώπων ε, εξαρθρώνοντας τις εγκληματικές ε, σπήρες και αντιμετωπίζονται στη δράση του. Σήμερα έχουμε ε, έχουμε σταματήσει τις, ε, αυτές τις ροές σε μεγάλο βαθμό και έχουμε φέρει ενώπιον της ε, δικαιοσύνης τους ηθήνοντες και έχουμε διασώσει ε, χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα. Όμως κάνουμε και άλλα πράγματα για να διαταράξουμε το έργο των εγκληματικών σπυρών συγκέντρωση, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών ε, σε σχέση με αυτά τα δίκτυα. Όλο ένα και περισσότερο αυτό μας βοηθάει να αναλύσουμε καλύτερα τον ρόλο που έχει το οργανωμένο έγκλημα σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση και τα μέσα για να διαταράξουμε αυτές τις ε, λειτουργίες. Η διακήρυξη της Μάλτας έδωσε νέα έμφαση στη συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου. Ενισχύουμε λοιπόν τη συνεργασία μας με τη Europol, τη Eurojust, τις Ιταλικές Αρχές, τον Frontex, με τον οποίο έχουμε πολύ στενή συνεργασία και έχουμε εντοπίσει τομείς όπου ενισχύουμε τις κοινέ μας προσπάθειες. Όπω ανέφερε και ο Επίτροπο Κίνγκ, η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο τη κοινή μα και συλλογική μα ανταπόκριση. Σύντομα, ε, συνυπογράψαμε μια συνεργασία με την Μάρκομ που είναι ε, φορέας του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της συνεργασίας. Είναι ένα πολύ καλό βήμα για να έχουμε μελλοντικά ένα νέο ε, πρόγραμμα πλαίσιο για τη συνεργασία και σε αυτόν τον τομέα και σε άλλους. 89% των μεταναστών που διέρχονται τη Μεσόγειο πέφτουν θύματα διακίνησης από τη Λιβύη και πρόκειται για μια ακτογραμμή που είναι μόνο 31 χιλιόμετρα. Επομένως, ε, βρισκόμαστε κοντά σε μια λύση. Πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο με τους reviews ε, φίλου μα και εταίρου μα για να του βοηθήσουμε και να σταματήσουμε τελικά κάθε μορφές ε, παράνομη διακίνηση και να σώσουμε ζωέ. Η επιχείρηση Σοφία έχει μας έχει δώσει πολύ καλές δομές κατάρτισης. Είμαστε ο μοναδικός οργανισμός που συμβάλλει στην υλοποίηση του εμπάργου όπλων του ΟΗΕ κατά της Λιβύης. Ευχαριστώ. Ε, muchas Σας ευχαριστώ, κύριε Φοντίνη. Μόλις έφτασε και κάθισε δίπλα μου ο Υπουργός Μετανάστευση και Δικαιοσύνη τη Σουηδία, ο κύριο Μόρχαν Γιώχανσον. Καλώ ήρθατε. Άρα θα δώσω πρώτα το λόγο στη συνάδελφο Αναγκόμε. Χωρί μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Ο κύριος λόγος για τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εσωτερική ασφάλεια σε μία διάσκεψη για τη μετανάστευση, η οποία είναι λίγο παράλογα οργανωμένη, ε, είναι όχι γιατί οι μετανάστες συνιστούν κίνδυνο, αλλά λόγω της ανεπάρκειας, της απόλυτης ανεπάρκειας των κυβερνήσεών μας στην ενσωμάτωση των μεταναστών. Και αυτό οδηγεί και στις, ε, στο να λεσμονούμε ορισμένοι ότι είναι ενδογενείς οι επιθέσεις. Βλέπουμε αντίστοιχα ως λόγο αυτών των επιθέσεων μεγάλες ε, περικοπές στις δυνάμεις ε, τήρησης του νόμου και ασφαλείας Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει διαλειτουργικότητα, εάν οι δυνάμει ασφαλεία δεν είναι σε θέση να παρακολουθούν τι δραστηριότητε εκείνων που ήδη είναι και καταγεγραμμένοι στα αρχεία ω πιθανοί τρομοκράτε, ε, χάνουμε ε, πολύ μεγάλο δυναμικό. Επίση, εάν δεν επενδύσουμε με τρόπου ασφαλού και νόμιμους ε, στην υποδοχή των προσφύγων, ουσιαστικά τροφοδοτούμε την διακίνηση, δίνουμε τους ανθρώπους αυτούς βορρά στους διακινητές και όπως είπε και ο Αντώνιο Κουτέρες, αυτή είναι τα πραγματικά θύματα της μετανάστευσης ε, με τα κέντρα κράτησης, hot spots στις χώρες μας ή στη Λιβύη ακόμη που είναι πραγματικά στρατόπεδα κράτησης όπως είπε και ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ εδώ μέσα στο κοινοβούλιο εχθές, εκπρόσωπος των ΗΠΑ στη Λιβύη με βασανισμούς, με παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων πάλι δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στη ρίζα τους και η ρίζα των προβλημάτων αυτών είναι όλες αυτές οι πολιτικές οι οποίες διαιωνίζουν την κλεπτοκρατία και δεν επιτρέπουν στις χώρες αυτές τις γειτονικές της Ευρώπης, στις χώρες Αφρικής δηλαδή, να σταθούν στα πόδια τους σε κράτο δικαίου. Και βεβαίως θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη ροή του χρήματο, όπως υπόθηκε και νωρίτερα. Πρέπει εμείς να μεριμνήσουμε στα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους και ό,τι οφείλουν να πράξουν για την πάταξη τη νομοποίησης παρανόμων εσόδων που τροφοδοτεί τρομοκρατία, γιατί αυτό δεν το πράττουν. Ευχαριστώ, Άννα, που υπερασπίζεσαι τη ιδέα σου, όπω πάντα, με τόση αποφασιστικότητα και τόση σαφήνεια. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο σε έναν άλλο συνάδελφο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, στον κύριο Κωνσταντίνο Καρβούνη. Καραγκούνη. Καραγκούνη, συγγνώμη. Πολύ επιγραμματικά κάποιε παρατηρήσει για το ζήτημα τη εσωτερική ασφάλεια, διότι επιτρέψτε μου να πω με όσα συμβαίνουν με τα τρομοκρατικά χτυπήματα, ε, απειλείται όχι μόνο η ασφάλειά μας, αλλά ο ίδιος ο τρόπος ζωής μας. Αναφέρθηκε νωρίτερα και συμφωνώ. Έχει γίνει σημαντική δουλειά τον τελευταίο καιρό, οδηγίες, κανονισμοί, το νέο χαρτοφυλάκιο για την ασφάλεια, η πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος έγκεν δεύτερης γενιάς, όπως και το δίκτυο RAN, το ETIAS, το ECTC και άλλα βεβαίως, ε, είναι πολύ σημαντικά βήματα. Όμως ας δούμε την πραγματικότητα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή συγκαταλέγεται στις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες με τον υψηλότερο αριθμό ετοιμάτων ασύλου. Πρέπει επιτέλους κάποια κράτη-μέλη να σταματήσουν να βλέπουν την κατάσταση κοντόφθαλμα και ωφελημιστικά και να συμφωνήσουμε όλοι σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό επιστροφών των μη δικαιούχων στις χώρες καταγωγής τους ή σε τρίτες χώρες. Το βάρος πρέπει να το αναλάβει η Ευρώπη συνολικά και όχι το κάθε κράτος χωριστά ώστε οι ιδιοκτικέ αρχές και οι αρχές ασφαλείας να κάνουν πολύ πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Πρέπει επίση η Ευρώπη να εξετάσει πιο αποφασιστικά το ενδεχόμενο δημιουργία κέντρων υποδοχής σε τρίτες χώρες, όπου θα γίνεται η επεξεργασία των ετοιμάτων ασύλου με ασφάλεια και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίω θα ελέγχονται πολύ πιο σωστά και έγκαιρα οι ροές από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Τέλος, θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών πληροφόρησης, συγκέντρωση και ομογενοποίηση των πληροφοριών τόσο στα κράτη-μέλη όσο και στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Δυστυχώς, και με αυτό κλείνω, σε πολλά κράτη-μέλη, όπως και στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας. Υπάρχουν κατακαιρματισμένες υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται σε ξεχωριστούς φορείς Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση και στα μέσα και σε προσωπικό και κυρίως κοινή στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφοι. Και τώρα θα δώσω το λόγο στου δύο τελευταίους ομιλητές. Γιατί κατεβαίνει όπου να είναι και ο πρόεδρος Ταγιάννη. Ο πρώτος είναι από το Πρωτοκαλικό Κοινοβούλιο, ο Αντώνιο Φιλίπε. Είναι ο πρώτο τελευταίο ομιλητή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τεράστιο θέμα, πολύ σημαντικό. Και είναι και ένα θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε. Αυτό σημαίνει συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και επαρκή μέσα. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα να προσθέσω δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας. Δεν πρέπει να θεωρηθούν εκ προημίου εγκληματίες. Το να αποδώσουμε αυτή την αρμοδιότητα στην αστυνομία είναι σαν να στιγματίζουμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Στην πραγματικότητα πρέπει να τους προστατεύσουμε. Επίσης, η ασφάλεια δεν πρέπει να δικαιολογεί τη δημιουργία ενός κράτους που θα έχει αιμονή με την ασφάλεια. Ε, Ενό αστυνομικού κράτου που θα ασχολείται συνέχεια με την ασφάλεια. Θα πρέπει να παντρέψουμε την ασφάλεια και την προστασία των ελευθεριών και δικαιωμάτων των πολιτών, όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από την εθνική του προέλευση και από τις σκεφτικές πεπιθήσει. Ευχαριστώ. Και εγώ σα ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Και τώρα, τελευταίος ομιλητή είναι ο Σιμών Θινκόφσκι από, την, ε, από το Κοινοβούλιο της Πολωνίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι λυπηρό που ακούσαμε με τόση υπομονή ε, τα κηρύγματα του, των κυρίων Γιούνκερ και Ταγιάννη, αλλά δεν είχαν εκείνη το χρόνο ε, να ακούσουν τι έχουν να πούν και εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, που σε τελική ανάλυση έχουν και αποφασιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική. Τώρα, η Πολωνία βεβαίως ε, και τηρεί και σέβεται την αρχή της αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά σύνορα και μάλιστα είναι τα ε, μεγαλύτερα εξωτερικά σύνορα από πλευράς χωρών, ε, πάνω από 1100 χιλιόμετρα. Ε, δαπανώνται τεράστια ποσά ε, για τον εξοπλισμό που είναι τεχνολογίας εχμής και με πάρα πολλούς ανθρώπινους πόρους επίσης. Έχουμε 118.000 ε, αφιχθέντες ε, στη Σέγγεν, αλλά 390 άτομα έλαβαν το καθεστώς του πρόσφυγα υπό τη Σύμβαση της Γενέβης και έτσι μπορούμε να πούμε ότι η Πολωνία όντως εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, Έχουμε αποστείλει πάνω από 400 αξιωματούχου για την προστασία των συνόρων ε, ε, του χώρου Σέγγεν στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Αλλά δεν θα συμφωνήσουμε στο ε, σύστημα επανακατάσταση γιατί θα, θα λύσει κανένα πρόβλημα. Αντιθέτω, θα μα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερε δυσκολίε σε ό,τι αφορά τον τομέα τη ασφάλεια. Θέλουμε να βοηθήσουμε του μετανάστε, αλλά δεν θα μα οδηγήσει η αρχή τη αλληλεγγύη για να μα δημιουργήσει προβλήματα. Ήθελα να σα πω το εξή. Αυτή η πολύ σημαντική συνάντηση υψηλού επίπεδου οργανώθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Ταγιάννη. Ο κύριος Ταγιάννης ε, ε, προσκάλεσε τους εθνικούς βουλευτές. Και αυτό που είπε στην ομιλία του, στην αρτήρια ομιλία του, μου φάνηκε πολύ σωστό, πολύ κέριο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους και σταματάω για μία στιγμή την ε, συνεδρίαση αυτή, γιατί τώρα θα πρέπει να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της ε, συνεδρίας αυτής. Σας ευχαριστώ όλους.